Σα Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. η προφορική ερώτηση σχετικά με την απλούστευση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ο κύριος Νίκολσον, ο ένας από τους τρεις ομιλητές, δεν είναι εδώ τώρα και έτσι θα απευθυνθώ πρώτα στον κύριο Ντες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Τσόλος. Χαίρομαι ιδιαίτερος που παρίσταστε εδώ σήμερα και θα μπορέσετε να απαντήσετε στην ερώτηση, διότι το, στις 18 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το κοινό ψήφισμα σχετικά με την απλούσευση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Βεβαίως μέχρι στιγμή αυτό το ψήφισμα δεν έχει εφαρμοστεί, αλλά θα παρακαλούσα κύριε Επίτροπε στη νέα ρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής να φροντίσετε οι απαιτήσει που περιλαμβάνονται σε αυτό το ψήφισμα να ληφθούν υπόψη διότι δι, δυστυχώς έρχομαι από μια συζήτηση με γεωργούς και πρέπει να σας πω ότι οι γεωργοί εξέφρασαν το φόβο ότι οι προτάσεις τις οποίες κάνατε στον πρώτο πυλώνα κύριε Επίτροπη δεν μειώνουν την ε, ε, γραφειοκρατία αντιθέτως τη διευρύνουν πάρα πολύ. Ε, κύριε Επίτροπε Τσόλος, δεν ευθύνεται για κάθε γραφειοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πολλές φορές ευθύνονται και τα κράτη-μέλη. Θα σας παρακαλούσα όμως από κοινού να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε αυτή την αναθεώρηση, κατά τρόπον ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν ε, λιγότερο γραφειοκρατικό βάρος, κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να αφοσιωθούμε στην ουσία, δηλαδή την παραγωγή τροφίμων και να μην χρειάζεται κάποιος ε, να διαβάσει ένα μακρύ κείμενο προτού μπορέσει να καλλιεργήσει το χωράφι του. Διότι υπάρχουν τόσες διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, ε, είναι ένα θέμα που δεν είναι τη δικιά σας αρμοδιότητα κύριε Επίτροπε αλλά θα μπορεί να γίνεται ο πρώτος Επίτροπος δεν ξέρω πότε θα αποσυρθείτε αλλά να πείτε ότι στη δικιά μου εποχή δεν αυξήθηκε η γραφειοκρατία μειώθηκε και γι' αυτό σας προτείνω να βρούμε από κοινού μία λύση για το πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Λιόν, ο δεύτερος Λάιον. Χαίρομαι που σας βλέπω κύριε Επίτροπε μαζί μας απόψε. Σαφέστατα η απλούστευση και εξαφάνιση της γραφειοκρατίας από την ΚΑΠ είναι βασικό βασικός στόχος γιατί πολλοί αγρότες στη Σκοτία είναι θυμωμένοι με τη γραφειοκρατία και την ε, δυσανάλογη, ε, τον δυσανάλογο μηχανισμό ποινών. Βεβαίως πρέπει να ελέγχονται τα χρήματα πως δαπανώνται, αλλά δεν υπάρχει αναλογικότητα στο σημερινό σύστημα κυρώσεων και στο επίπεδο των κρατών μελών αλλά και στο επίπεδο του ε, ατομικού αγρότη. Και είναι κάτι που πρέπει να το λύσετε με τη μεταρρύθμιση. Τιμωρούνται για μικρά λάθη αγρότες στην Σκοτία και μάλιστα με μεγάλες ε, κυρώσεις, οικονομικές κυρώσεις. Οι ποινές διανέμονται ευρύτατα ε, ε, η σκοτική κυβέρνηση ε, θεωρεί ότι εσείς φταίτε κύριε Επιτροπέ για το σύστημα με το οποίο κλείνουν οι επιθεωρήσεις και επιβάλλονται οι ποινές. Μια εξήγηση μπορεί να είναι ότι οι επιθεωρητές της Κομισιόν έρχονται έρχονται τακτικά στη Σκοτία τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και μπορεί ε, η κυβέρνηση της Σκοτίας να έχει τρομοκρατηθεί από τις δρακόντιες ποινές που επιβάλλονται τους τελευταίους τρεις-τέσσερις μήνες. Ε, ανησυχούν όλοι ότι μπορεί τα πράγματα να μην είναι άψογα όταν θα φτάσουν οι επιθεωρητές σας. Αλλά ας κοιτάξουμε ε, και τι γίνεται με τους συναδέλφους στη Βόρεια Ιρλανδία και σίγουρα ο ο Νίκολσον θα πει δύο λόγια γι' αυτό. Για να δούμε τι γίνεται με τη δικιά τους κυβέρνηση. Έχουν αντιμετωπίσει τεράστια μάχη για την παρερμηνία ορισμένων μέτρων ε, και αυτά συναρτίζονται με τη Σκοτία. Λοιπόν, κύριε Επίτροπε, μπορείτε να εξηγήσετε αν πραγματικά η Κομισιό είναι υπεύθυνη για το δρακόντιο καθεστώς που επιβάλλεται στη Σκοτία και ε, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι είναι της Κομισιόν οι επιθεωρήσεις που έγιναν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και επέβαλαν τόσο δρακόντιες ποινές. Κύριο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ. Συγγνώμη που δεν ήμουν στη θέση μου ότι μου δώσατε αρχικά το λόγο. Δεν το συνηθίζω αυτό. Η Ολομέλεια σίγουρα γνωρίζει ότι ο συνάδελφος, η έκθεση του συναδέλφου Άστον εγκρίθηκε ε, το περασμένο Μάιο για να καταργηθεί η γραφειοκρατία που επιβάλλεται στους Ευρωπαίους αγρότες και που έχει γίνει πολύ επιβαρυντική και παρεμποδίζει αν θέλετε την εξέλιξη ε, αντί να καλλιεργούν υποβάλλονται στη γραφειοκρατία η μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ πρέπει να ευθυγραμμιστεί σωστά Φοβάμαι λοιπόν ότι δεν οδηγούμεθα όμως αυτό. Οδηγού, ε, μας πάνε σε περισσότερη γραφειοκρατία. Και όταν μιλάμε για το πρασίνισμα του τρίτου πυλώνα, τι προσπαθείτε να πείτε. Ουσιαστικά λέτε περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότερα χαρτιά για τον αγρότη, περισσότερες επιθεωρήσεις και δεν είναι αυτό που θέλουν. Θέλουμε μία επιθεώρηση κάθε, ε, κάθε εκμετάλλευσης και αυτό πρέπει να επαρκεί ε, έχετε την πολλαπλή συμμόρφωση αυτή τη στιγμή. Δεν χρειαζόσαστε Κομισιόν τίποτα παραπάνω σε σχέση με τους ελέγχους. Και ε, κάνω έκκληση εκ μέρους όλων αυτών που προσπαθούν να παράγουν. Μιλάμε για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη. Μα σας την έχουμε δώσει αυτή την ασφάλεια. Αφήστε τους αγρότες να παράγουν. Θα ήθελα επίσης να συνεχίσω από αυτό που είπε ο κύριος Λάιονς. Οι αγρότες στη Βόρεια Ιρλανδία έχουν ποινές 60 εκατομμύρια ευρώ. Και κανένας δεν αμφισβητεί ότι οι χάρτες ε, που δημιουργήθηκαν πριν από χρόνια είναι ε, τέλειοι. Δεν είναι. Ε, δεν ξέρω αν είναι καλύτεροι στην Ιταλία ή στη, από την άλλη πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας. Αλλά γιατί επιβάλλονται αυτά τα δρακόντια μέτρα όταν δεν χρειάζονται και το μόνο που θέλουν οι αγρότες είναι να φτιάξουν, να παράγουν καλά τρόφιμα. Πρόεδρος. Ε, Επίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε τις ερωτήσεις. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να δώσω κάποια, κάποιες απαντήσεις πρώτα απ' όλα στην γραπτή σας ερώτηση όσον αφορά την απλούστευση. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό όπως το έχω πει από τότε που ανέλαβα επίτροπος. Είναι ένα θέμα που το λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη στον κανονισμό που σχεδιάζουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω το πρώτο στοιχείο της ερώτησής σας. Τι έχουμε κάνει προς το παρόν για να απλουστεύσουμε το βίο των αγροτών. Αν πάρουμε το τι έγινε τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι η Κομισιό ήδη απλούστευσε σημαντικά. Ήδη έχει εφαρμόσει μέτρα για την απλούστευση Τον ε, Μάρτιο του 2009 είχαμε την ανακοίνωση για την ε, απλούστευση της ΚΑΠ. Και αυτή η ανακοίνωση προωθεί τις δραστηριότητες των τελευταίων ετών και δίνει ενδείξεις σε σχέση με τη μείωση του διοικητικού βάρους που επετεύθη. Δεν θα τα επαναλάβω όλα όσα εμπεριέχονται σε αυτή την ανακοίνωση, θα σας δώσω παραδείγματα. Το 2007 έχουμε τον κανονισμό του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των γεωργικών Πράγμα το οποίο οδήγησε σε σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας μέσα στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την ΚΑΠ. Λόγω του τεχνικού χαρακτήρα η οργάνωση της ενιαίας αγοράς δεν τροποποίησε αν θέλετε τη βάση αλλά εξαρμόνισε τις διατάξεις ώστε η ΚΑΠ να είναι πιο εύκολη στην εφαρμογή της. Η απλούστευση επίσης ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησε στον απολογισμό της Κομισιόν ε, και αν θέλετε τον κανονισμό του 2009 που διευκολύνει τις ενιαίες ενισχύσεις ε, και αλλάζει την ΚΑΠ του 2003. Έχουμε πρόοδο λοιπόν στον αγροτικό τομέα. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στη μείωση του διοικητικού βάρους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα προγράμματα ε, οδηγήθηκαν σε πολλαπλές αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις λοιπόν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κατά 36% είχαμε μείωση του γραφειοκρατικού βάρους υπερβαίνοντας το στόχο του 25%. Ο προκάτοχός μου επίσης απάντησε στον κατάλογο των 35 απλουστεύσεων που είχαν υποβληθεί τον Απρίλιο του 2009. Ένα κομμάτι αυτών των απλουστεύσεων είχαν εφαρμοστεί στο τέλος του 2009, αρχή 2010. Το δεύτερο μέρος εμπεριέχεται όσον αφορά, στο νέο πακέτο της Κομισιόν όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενιαία ανίσχυση. Το έχουμε υποβάλει στο Κοινοβούλιο. Για το δεύτερο πυλώνα έχουμε ε, ξεκινήσει μία μελέτη για την ανάπτυξη τη γεωργική με επικέντρωση σε δύο μέτρα. Το αγροπεριβάλλον και τον εξυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών θα χρησιμοποιηθούν για την ΚΑΠ μετά το 2013. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι το πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει και την διαμονή ενός στελέχους σε εκμεταλλεύσεις αγροτικές, το Harvest Experience όπως αποκαλείται, μας βοηθάει επίσης να έρθουμε σε άμεση επαφή με, τον το αγροτικό περιβάλλον. Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο της ερώτησής σας, πώς η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τις συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου για μετά το 2013, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ενδιαφερόμεθα πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις αναλύσεις που έχουν ήδη γίνει για να απλουστεύσουμε και θα προχωρήσουμε σε προτάσεις που δεν οδηγούν σε περισσότερη γραφειοκρατία, αλλά περισσότερη, σε περισσότερη διασφάλιση για τον ενδιαφερόμενο και για την καλή χρήση των χρημάτων και των κοντιλίων. Είμαι ανοιχτό για οποιαδήποτε τεχνική πρόταση που θα κάνετε. Αρχές Δεκεμβρίου θα έρθω ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Και εκεί με ρωτούν τι έχει κάνει η Κομισιό για να εξασφαλίσει ότι το δημόσιο χρήμα χρησιμοποιείται σωστά. Η Κομισιό εφαρμόζει κανονισμούς που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο και με τη γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν προσθέτουμε εμείς διοικητικό βάρος, εμείς η Κομισιόν δηλαδή εφαρμόζουμε τους κανονισμούς του Συμβουλίου που είναι ήδη ενισχύ. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι στο μέλλον δεν θα έρθουμε με προτάσεις που θα περιπλέκουν τα πράγματα. Θα καταστήσουμε την ΚΑΠ πιο αξιόπιστη στο περιεχόμενό της. Για τον αγρότη, ο βασικός του ρόλο είναι η παραγωγή. Και ο ίδιος αγρότης εργάζεται με τους φυσικούς πόρους και εξ αυτής της ε, δραστηριότητας του δίνονται κονδύλια της ΚΑΠ. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα μετά το 2013. Προσπαθώ να σας ενημερώσω ότι εκπαραλλήλουμε ένα νομοθετικό πακέτο για την ΚΑΠ μετά το 2013. Ε, αποφάσισα να δημιουργήσω ένα, μια ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου με τα κράτη-μέλη για να προετοιμάσουμε το νομοθετικό πακέτο ώστε να εξασφαλίσουμε να μην προσθέσει αυτό το πακέτο γραφειοκρατία. Όπως είπε ο Λάιον, Πολύ συχνά η γραφειοκρατία που βρίσκει τον αγρότη στο ε, κάμπο του, στο χωράφι του, δεν οφείλεται στην Κομισιόν. Έχουμε καμιά φορά εφαρμογές διαφορετικές από χώρα σε χώρα βάσει της εθνικής διοίκησης κάθε μίας. Η Κομισιόν έχει ήδη απλουστεύσει, αλλά θα πρέπει να απλουστευτούν και οι διαδικασίες στο κράτος μέλος. Ε, όσον αφορά την ερώτηση του George Lyons για τη Σκωτία. Εδώ τηρεί η Κομισιόν τους κανονισμούς και όσοι αγρότες δεν συμμορφώνεται με την πολλαπλή συμμόρφωση υπάρχουν ποινές οι οποίες εφαρμόζονται όχι μόνο στη Σκοτία και στη Βόρεια ε, Ιρλανδία αλλά σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένας κανονισμός που αν δεν εφαρμόζεται δεν είμαστε πλέον εμείς αξιόπιστοι όσον αφορά την νομοθεσία την ευρωπαϊκή. Η πολλαπλή συμμόρφωση δεν είναι κανόνας που προστίθεται ένα κράτος μέλος και ένα άλλο, είναι η κοινοτική νομοθεσία, η ενωσιακή νομοθεσία. Ε, η κυβέρνηση θα λάβει από την Κομισιόν στην αρχή Δεκεμβρίου τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα περνάμε στους ομιλητές εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την οθόνη. Ο κύριος Νίκολσον έχει μία, ο κύριος Down, έχει μιλήσει, ο κύριος Downtown Η κυρία Downtown θα μιλήσει, με συγχωρείτε, για δύο λεπτά εκ μέρους του ΕΛΚ. Κύριε Επίτροπε, είστε απόλυτος γνώστης της γαλλικής γλώσσας, γνωρίζετε τη χώρα μου. Αλλά στην ε, χώρα μου έχουμε μία έκφραση την Αγλυζία. Λοιπόν, υπάρχει όπως και στην Αρλεζία εδώ μία διπλή μορφή. Έχουμε αφενός τους φακέλους όπου ζητεί, βοήθεια. Και μετά έχουμε και τις δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την κοντινσιοναλιτέ. Ας πούμε θα πρέπει, πρέπει οι αγρότες να λένε πόση κοπριά φόρτωσαν στο φορτηγό, πόσο λίπασμα ρίξανε, τι κάνανε και τι δεν κάνανε. Και άμα δεν τα αναφέρουν όλα αυτά, τότε πέφτουν πρόστιμα. Λοιπόν, όταν παρουσιάσατε το σχέδιο για την μελλοντική ΠΑΚ, μιλήσατε για σχέδια ολοκλήρωσης τα οποία ζητούν μέτρα όπως είναι οι κυκλωτικές καλλιέργειες για παράδειγμα όπου μπορεί είναι μέτρα τα οποία και ελέγξιμα από τις υπηρεσίες της Κομισιόν και εφαρμόσιμα για τους αγρότες. Μετά αναφέρατε και τι εμπίπτει στα κράτη-μέλη. Πριν πάνε οι ελεγκτές της Κομισιόν στους χωρικούς, πηγαίνουν πρώτα στα κράτη-μέλη και προσπαθούν να δουν τι δεν λειτουργεί. Δεν θα μπορούσαμε όμως αυτούς τους ελεγκτές να τους προωθήσουμε λίγο στην αποστολή τους και να μπορέσουν να συγκρατήσουν τα κράτη όταν παρατραβάνε το σκηνή στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και επιβάλλουν τεράστιες υποχρεώσεις στους γιοργούς. Έτσι θα βελτιώνατε και την εικόνα της Ευρώπης στους πολίτες. Ο κύριος Κάπουλα Σάντος για δύο λεπτά. Εδώ και χρόνια τα φωνάζουμε όλα αυτά. Αλλά ακόμη δεν έχουμε προσεγγίσει τίποτα παρά τις ε, συνεχείς προσπάθειες της Κομισιόν. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες η απλούστευση δεν μπορεί να θεωρείται ως οποιοδήποτε άνοιγμα στην ε, κατάργηση των ελέγχων ε, και στην χαλαρότητα δεν πρέπει με τίποτα να χαλαρώσουμε εμείς τη διαφάνεια με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ έχουμε μια τεράστια ευκαιρία για να προσεγγίσουμε το στόχο της διαφάνειας αλλά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε όμως απλούστευση αν δεν απλουστεύσουμε και την ίδια τη δομή της ΚΑΠ. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν εκφράστηκε η σοσιαλιστική ομάδα τον προηγούμενο Απρίλιο. Δημοσιεύσαμε τότε ένα έγγραφο για την αναδιοργάνωση των δύο πυλώνων και διαπιστώνουμε με μεγάλη ικανοποίηση ότι η Κομισιόν έλαβε υπόψη τις ορισμένες από τις προτάσεις μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν καταλαβαίνουμε πώς μετά από τον διαχωρισμό με, με κριτήρια για την προστασία του περιβάλλοντος, άμεσες πληρωμές, ε, ε αγροπεριβαλλοντικά μέσα, ε, βοήθειες για τις λιγότερες, ε, για τις πιο συγγνώμη, περιοχές, γιατί έχουμε διαφορετικά διαφοροποιημένες πληρωμές πάντα γιατί το, το ενιαίο σύστημα δεν λειτουργεί και με δυσκολία εμείς ε, μπορούμε να καταλάβουμε όλα αυτά τα ωραία λόγια για την απλούστευση και μετά βέβαια είναι αυτοί που αντιστέκονται περισσότερο για τη νέα δομή της ΚΑΠ. Εμείς επενούμε τις εργασίες του Επιτρόπου Τσόλος, περιμένουμε άμεσες προτάσεις και ευχόμαστε όλοι όσοι είναι υπέρ της απλούστευσης ας το αποδείξουν με συγκεκριμένες πράξεις στη συζήτησή μας για την ΚΑΠ. Κυρία Ράιμερς, για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η μείωση της γραφειοκρατίας και ε, η ε, απλοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτη στι προτεραιότητες για τους ευρωβουλευτές για να μπορέσουμε ε, να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα των φορολογουμένων και να γίνουμε αποδεκτοί από τους πολίτες. Γι' αυτό και είναι βασικό στο γεωργικό τομέα να μπορέσουν να να φτάσουν αυτές οι δυνατότητες εις ε, τους γεωργούς για να μπορούν να παράγουν τρόφιμα και θα πρέπει εις ε, μια εποχή που μειώνεται ο προπολογισμό να φροντίσουμε ε, να υπάρξουν κανονισμοί οι οποίοι να μπορούν να εφαρμοστούν και να μην παραμένουν στο ράφι. Άλλωστε πρέπει να φροντίσουμε οι κυρώσεις να είναι αντίστοιχες με τις παραβάσεις μία αηφόρος πολιτική ε, χαρακτηρίζεται με προστιθέμενη αξία και όχι με κυρώσεις και τιμωρία γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα στους πολίτες και στους γεωργούς για να μπορέσουν να καλύψουν τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν θα μιλήσουμε για την μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική και να φροντίσουμε με μεγάλη προσοχή να μην υπάρχει επικάλυψη των ελέγχων, των ε, διατυπώσεων και να υπάρξει γραφειοκρατία μόνο όταν ουσιαστικά υπάρχει προστιθέμενη αξία και για τη διαχείριση αλλά και για τον ε, Γεωργό για να συνεργαστούμε και να μην αντικρουόμαστε κατά την ε, εξέλιξη αυτή. Ο κύριος Σμίθ για 1,5 λεπτό εν ονόμα των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των Πρασίνων και θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο που είναι εδώ απόψε και θα ήθελα να συγχαρώ συναδέλφους και τον κύριο Ashworth ειδικότερα για το ψήφισμα. Αναφέρομαι στις παραγράφους 52 και 53 όσον αφορά την διαφάνεια των ποινών εκτός από το εσωτερικό μας έχουμε πρόβλημα στη Σκοτία και σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά τη διαφάνεια για τους αγρότες και την πολλαπλή συμμόρφωση. Για να προχωρήσουμε χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια ως προς το τι απαιτείται και τι περιμένουμε από τους αγρότες. Χρειαζόμαστε ακόμη να δούμε καλύτερη κατανόηση και ευελιξία. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε κανονισμούς που έχουν γραφτεί, αλλά ελπίζουμε ότι θα τους ξαναγράψετε. Αυτό να μένουμε. Υπάρχει διαφορά μεταξύ ατυχήματος και απάτης. Και, και στις δύο περιπτώσεις μεταχειρίζεσαι τους αγρότες με τον ίδιο τρόπο. Στην παραγράφο 66 θα ήθελα μια ένδειξη από εσά κύριε Επίτροπε σχετικά ε, σχετικά με το πώς βλέπετε την περίπτωση των αγροτών και την πολλαπλή συμμόρφωση και την αναγνώριση την ηλεκτρονική και την αναβολή της για τρία χρόνια. Θα προσπαθούμε να λειτουργήσουν όλα αυτά. Ξέρουμε ότι είσαστε ευέλικτες. Ε, θα θέλαμε να μας διαβεβαιώσετε ότι θα έχουμε μια μεταβατική περίοδο τριών ετών. Ο κύριος Άσχουρθ, εκ μέρους της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εγώ έγραψα την αρχική έκθεση και σε αυτή την έκθεση μίλησα για τις προκλήσεις για τη Γεωργία και τόνισα τους τρόπους με τους οποίους η ΚΑΠ πρέπει να μεταβληθεί για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Την έκθεση επέστειρα την προσοχή στο γεγονός ότι πολλοί τομείς γεωργίας και η κτηνοτροφία ειδικότερα αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες και υπάρχει επίγουσα ανάγκη να μειώσουμε το βάρος όσον αφορά τον χρόνο και το κόστος για τους αγρότες λόγω μην απαραίτητων όρων και ρυθμίσεων. Οι ποινές είναι δυσανάλογες πολύ συχνά, θα έλεγα και άδικες καμιά φορά αναφέρομαι στην ανάγκη αξιολόγησης των συνεπειών, των επιπτώσεων, την εναρμόνιση των κανόνων και πρότεινα ακόμη ότι η αυτορύθμιση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επιτυχημένα στη Γεωργία. Και θέλω και μία μεταβολή του όλου πολιτισμού γύρω από την ΚΑΠ. Βεβαίως και καταλαβαίνω την ανάγκη διαχειριστικής ακαιρεότητας. Αλλά το ελεγκτικό συνέδριο έχει καταδείξει ότι πολλές φορές οι υπερβολικές περιπλοκές είναι η αιτία των προβλημάτων. Η διαχείριση και η ερμηνεία των κανονισμών διαφέρουν πολύ από μία χώρα σε μια άλλη. Αφού έγραψα την έκθεση, χαίρομαι που διαπίστωσα ότι πολλές κυβερνήσεις και σημαντικές γεωργικές οργανώσεις επιδιώκουν την απλούστευση. Τώρα κύριε Επίτροπε που συζητάμε την ΚΑΠ και τη μεταρρύθμισή της είναι ο καλύτερος χρόνος για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε το κλάδο χωρίς να τον παρεμποδίζουμε ε, με κόστος και γραφειοκρατία που δεν είναι απαραίτητα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε κάνει βήματα πρόοδου αλλά ανησυχώ που δεν έχει περάσει το μήνυμά σας στους αγρότες. Σας ευχαριστώ. Θα το πω μία φορά είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Έχουμε πολλούς που ζητούν να μιλήσουν για ένα λεπτό σύμφωνα με τη διαδικασία Catch the Eye και σας παρακαλώ πάρα πολύ να τηρήσετε το χρόνο ομιλίας γιατί αλλιώς δεν θα τελειώσουμε τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Φερέρα τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον περασμένο Μάιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα ψήφισμα για την απλούστευση της ΚΑΠ. Και είχαμε πει τότε ότι η απλούστευση δεν σημαίνει λιγότερη υποστήριξη προς, τους γεωργούς, ούτε θα έπρεπε να καταργήσει τις ε, κοινέ οργανώσεις αγοράς. Πέρασαν έξι μήνες τώρα από αυτό το ψήφισμα και παραμένουν πάντα σοβαρά, σοβαρές ανησυχίες ε, οι οποίες εντείνονται με την πρόσφατη ανακοίνωση της ε, Κομισιόν. ή παραδοσιακές μέθοδοι διαχείρισης των αγορών, δημόσιες πανεμβάσεις κτλ. δεν μπορούν να καταργηθούν μέσα από το επιχείρημα της απλούστευσης της ΚΑΠ διότι αυτό θα οδηγούσε σε πολλές χώρες την καταστροφή των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στην ΚΑΠ θετικά και απαραίτητα. Για παράδειγμα πώς να αλλάξουμε το σύστημα των κυρώσεων κυρίως ε, όταν αυτές αφορούν παραβιάσεις οι οποίες δεν είναι ευθύνη των παραγωγών. Υπάρχουν ε, αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην διαπίστωση των ε, και, και ταυτοποίηση των ζώων, αλλά οι περισσότεροι όμως είναι μικρομεσαίοι γεωργοί. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μία τροποποίηση που να ενισχύει τα μέσα παρέμβασης που να εγγυάται δίκαιες ε, τιμές ε, στην, ε, για την παραγωγή με την εγγύηση για κάθε χώρα όπως το δικαίωμα στην παραγωγή καταξιώνοντας την αρχή των ενισχύσεων για να ξεπεραστούν οι σημερινές ανισορροπίες μεταξύ χωρών και παραγωγών. Κύριε Επίτροπε, με μεγάλες ανησυχίες εμείς διαπιστώνουμε αυτές τις προτάσεις, αυτή την παρεμβατικότητα της Κομισιόν και τις προτάσεις της. Αυτή η πολιτική δεν έχει φέρει μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους μικρούς, μισέους γεωργούς, εγγυόμενοι μεγαλύτερα εισοδήματα και διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των διαφόρων περιφερειών της Ένωσης. Θα πρέπει οι μικρομεσαίοι γεωργοί να συνεχίσουν να παράγουν. Σε αυτήν την απλούστευση που προτείνεται σήμερα λέμε όχι. Ο κύριος Μπάφτον για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η ε, έκθεση για την αναθεώρηση της κοινή γεωργικής προοπτικής ε, τονίζει τη δεύτερη εναλλακτική λύση και υποθέτω ότι αυτήν επιλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε την κοινή γεωργική πολιτική προτού βελτιωθούν οι προτάσεις, προτού υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την πολλαπλή πολλαπλή συμμόρφωση διότι υπάρχουν ε, μικρές ε, εκμεταλλεύσεις και δεν έχουμε τρόπο να αξιολογήσουμε την ε, απόδοσή τους. Οι δύο πυλώνες δεν αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο και τα μικρά αγροκτήματα απέχουν από την παραγωγή για να μπορέσουν να επωφεληθούν από την κοινή γεωργική πολιτική ο στόχος μας είναι να υπάρξει διατροφική ασφάλεια και ανταπόκριση εις την ζήτηση ε, διεθνώς τροφίμων αλλά δεν βλέπω να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας και έχουμε υποχρεώσεις στο διεθνές εμπόριο. Η συμμετοχή μας στη γεωργία έχει μειωθεί ενώ έχει αυξηθεί η γραφειοκρατία μας. Οι συμφωνίες με το Μερκοσούρ και οι εισαγωγές μειώνουν τις δυνατότητες των Ευρωπαίων γεωργών να πωλήσουν τα προϊόντα τους σε μία δίκαιη τιμή και πρέπει να σέβονται διάφορους, διάφορες επιταγές ε, περιβαλλοντολογικές και άλλες ενώ τα εισαγόμενα προϊόντα δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ανεξάρτητο μέλος η κυρία Μορβάη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πολύ δημοφιλής στους μικρούς γεωργούς διότι ε, μεγάλα ποσοστά της αγοράς χρειάστηκε να απεμποληθούν για να μπορέσουμε ε, να ε, να καλύψουμε τις επιδοτήσεις των γεωργών. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, επιβαρύνσεις για τους Ούγγρους γεωργούς και πολλά εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν ε, στην ε, εξάσκηση των δραστηριοτήτων τους. Υπάρχει και ένας άλλος βασικός παράγων στην Ουγγαρία που προέρχεται από τη σοσιαλιστική εποχή οπότε ορισμένοι κρατικοί λειτουργοί θεωρούσαν ότι δεν χρειαζόταν να βοηθήσουν τους γεωργούς αλλά ότι οι γεωργοί ε, υπάρχουν για, το δικό τους, για να βοηθήσουν αυτούς. Ε, πράγμα το οποίο ε, δυσχεραίνει τη θέση των γεωργών και την επιβίωσή τους διότι επιβαρύνονται υπερβολικά με γραφειοκρατικούς κανονισμούς και οι γεωργοί συνέχεια παραπονούνται. Παραδείγματο χάρη, ορισμένοι από αυτούς δεν δέχονται ε, να ε, λάβουν πληρωμές από τον δεύτερο πυλώνα και ε, είναι ένα είδος Παραδείγματο χάρη να αναφέρω ότι ε, πρόσφεραν κάτι κρακεράκια τα οποία όμως δεν είχαν τιμολογηθεί σωστά και ηρωνεύτηκαν οι γεωργοί ότι δεν χρειαζόταν η τιμολόγηση αυτή. Ε, είναι όμως ε, αυτά όλα αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προσφέρει και τις επιδοτήσεις πρέπει να φροντίσει ε, για την επίλυση των προβλημάτων. Τώρα ανεξάρτητοι ομιλητές, ο κύριος Νικολέσκου πρώτα για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, καταρχήν να ευχαριστήσω για την δέσμευση της Κομισιόν στη δήλωσή της στο πλαίσιο δηλαδή της συνέχισης της απλούστευσης της ΚΑΠ. Όσο το δυνατόν πιο γραφειοκρατία έχουμε, τόσο λιγότερο η παραγωγικότητα έχουμε. Πρέπει λοιπόν να μεταρρυθμίσουμε την ΚΑΠ για να την απλουστεύσουμε. Τώρα, ε, πρέπει να σας θυμίσω το ψήφισμα που ήδη έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απλούστευση. Ο συνάδελφος Δαλτά μίλησε για την ε, γραφειοκρατική υπερβολή ορισμένων κρατών. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να την καταπολεμήσουμε όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να ορίσουμε ένα ανώτατο επίπεδο γραφειοκρατίας που, ένα όριο που δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί. Διότι εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει τρεις υπογραφές για ένα έγγραφο, στα εθνικά κράτη πολλές φορές ζητάνε πέντε. Πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν όλη τη χαρτούρα που είναι η απολύτως απαραίτητη. Πρέπει επίσης να ε, κοινοποιήσουμε ε, ε, την πληροφόρηση προς τους δικαιούχους διότι η απλούστευση συνδέεται με την διαφάνεια και εποφελούμε εδώ από την παρουσία του Επιτρόπου για να πω το εξής λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους δικιούχους των, αγροτικών επιδοτήσεων, τι σκοπό έχει η Κομισιόν, τι συνέχεια θα δώσει ο κύριος Ταραμπέλα Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ όπως ο συνάδελφος Νικολέσκου χαιρετίζω την προσπάθεια της Κομισιόν ε, για την απλούστευση, αλλά ανησυχώ όμως και για τη συνέχεια της έκθεσης ε, του συναδέλφου Σαρά για την ε, απλούστευση. Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη συγκυρία σήμερα των γεωργών μας, θα έπρεπε οι ΚΑΠ εν ώψη του 2013 να συγκεντρωθούν στο βασικό του στόχο, δηλαδή στην παραγωγή σίγουρων ασφαλών τροφίμων και ποιότητας και να παράγουν μη εμπορικά αγαθά, κοινά αγαθά. Θα πρέπει να περιορίσουμε την άχρηστη νομοθεσία και οι αγρότες από τις 27 χώρες θα πρέπει να μάθουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους αλλά και ποια είναι και τα δικαιώματά τους. Χρειάζεται λοιπόν μια κάπα με μεγαλύτερη αλληλεπίδραση. Ε, οι γεωργοί μας θεωρούν πολλές φορές τον παγκόσμιο ανταγωνισμό ως μοιραίο και μετά από τις ε, κρίσεις, τις τροφιμικές κρίσεις που γνωρίσαμε, θα πρέπει να βελτιώσουμε τις επαφές μας με τους γεωργούς, να δούμε τι γίνεται επί τόπου, να διεκδικήσουμε δίκαιες τιμές και δίκαιες τιμές και για τους καταναλωτές. Και να αναφέρω εδώ και τον Μποντλέρο, που, ο οποίος έλεγε ότι το υπέρτατο αγαθό για τη διάκριση είναι η απλούστευση. Θα έπρεπε λοιπόν και η Κομισιόν να πράξει το ίδιο μποντελεριανό σχήμα για να το πετύχει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη. Για μένα το πιο ενδιαφέρον ή σε, την, ε, ε, σε αυτό το ψήφισμα είναι ε, η γραμμή όπου λέγεται ότι πρέπει να αξιολογηθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος για να μπορέσουμε να έχουμε ένα βάρος αντίστοιχο με το στόχο που επιζητούμε συζητούμε. Μπορείτε να διεσμευτείτε κύριε Επίτροπε ότι θα ε, καλυφθούν αυτές οι προϋποθέσεις για την επόμενη κοινή γεωργική πολιτική του 2013 ότι θα, υπάρχει, ε, ε, θα υπάρχουν τρόφιμα ποιοτικά και καλής τιμής ότι θα μπορέσουμε να έχουμε πιο πράσινη ανάπτυξη, να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον, να υπάρχει βιοπικιλότης, να υπάρχει και ευημερία των ζώων, να καλύπτεται η πολλαπλή συμμόφωση και ε, να καλύπτονται και οι προδιαγραφές. Να υπάρχει σωστή ε, σειρά στην διατροφική αλυσίδα να ενταγωνιζόμαστε τις εισαγωγές και με μειωμένο προπολογισμό. Σας ευχαριστώ αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σας έδωσα πάρα πολλά επιχειρήματα για τις επόμενες συζητήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, Ε, πρέπει να μειώσουμε την υπερβολική γραφειοκρατία. Αυτή είναι η βασική απέτηση. Διότι οι γεωργοί χρειάζονται χρόνο για να μπορέσουν να ασχοληθούν με, ε, ε, την εργασία του στην ουσιαστική, δηλαδή τις καλλιέργειές τους και τα ζώα. Πρέπει λοιπόν να απλοποιήσουμε την κοινή γεωργική πολιτική όπως είχαμε δεσμευτεί το 2005 ότι θα μειωνόταν η γραφειοκρατία κατά 5% στο 2012. Βλέπουμε ε, κάποια αποτελέσματα αλλά δεν ε, καλύπτεται το κενό μεταξύ των κρατών μελών και δεν υπάρχουν ε, αρκετά αυτά αποτελέσματα. Η κοινή γεωργική πολιτική χρειάζεται ένα ευέλικτο πλαίσιο και θα πρέπει συγχρόνως να μειώσουμε και τους κινδύνους κατά τρόπον ώστε να επιτύχουμε πραγματική ποικιλία η απλοποίηση αυτή θα πρέπει να ε, ισοσκελίζεται και ε, με την, ε, με την αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, θα ήθελα να επανέλθουμε σε ένα σημαντικό θέμα. Τους τελευταίους μήνες έχουμε, έχω κάνει ορισμένες συναντήσεις με αγρότες στη Βόρεια Ιρλανδία. Κάθε φορά ζητάω τους αγρότες να μου μιλήσουν για τις βασικές αλλαγές που θέλουν στο τομέα τους. Τεράστια σημασία είναι η μείωση της γραφειοκρατίας που θεωρείται ότι επιβαρύνει σε κόστος και σε χρόνο ο όγκος της γραφειοκρατίας και η λεπτομέρεια που απαιτείται έχει δημιουργήσει μεγάλο βάρος για τους αγρόστες και ανησυχίες για ποινές. Πρόσφατα συναντήθηκα και με τους προέδρους ομάδων τοπικών που εφαρμόζουν το γεωργικό πρόγραμμα στη Βόρεια Ιρλανδία. Και εκείνοι μιλούν για τη μεγάλη επιβάρυνση των επιθεωρήσεων πράγμα που έχει οδηγήσει σε εγκαταλείψει. Βεβαίω απαιτείται λογοδοσία για τα χρήματα των φορολογούμενων, όμως η γραφειοκρατία παρεμποδίζει το πρόγραμμα και παρεμποδίζει τη συμμετοχή ανθρώπων που επρόκειτο να βοηθήσει. Ευχαριστώ κυρία Ζάμπου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπο. Πολύ συχνά μιλούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την απλούστευση της ΚΑΠ. Οι αγρότες μας όμως διαμαρτύρονται συνεχώς για τα διοικητικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ναι, όταν πρέπει να επιδιώξουν την ενισχύσει τους. Η Κομισιόν δεν είναι η μόνη που πρέπει να λάβει μέτρα και τα κράτη-μέλη πρέπει να το πράξουν. Πιστεύω ότι είναι ουσιαστικό η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη να γίνεται κατά τρόπο που να μην αποθαρρύνει τους γεωργούς. Πολλοί γεωργοί της χώρας μου διαμαρτύρονται διότι δεν είναι ενημερωμένοι και ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο να πείσει οποιονδήποτε να γίνει γεωργός σήμερα γιατί είναι κατατρομαγμένος με τη ε, γραφειοκρατία. Σας παρακαλώ λοιπόν η Κομισιόν να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη ώστε να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τη σημερινή τεχνολογία, να ενημερώσουν τους γεωργούς και να τους βοηθήσουν για να μειωθεί η γραφειοκρατία. Ελπίζω ότι η νέα ΚΑΠ θα είναι απλούστερη, διαφανέστερη και δικαιότερη. Ο κύριος Μίλντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε εδώ και καιρό σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο μιλάμε, για την απλούστευση της γραφειοκρατίας. Η Κομισιό ε, συνέστησε μια ομάδα εργασίας από τα στελέχη τα οποία πρέπει να φροντίσουν ώστε οι νομοθετικές ρυθμίσεις να μην είναι υπερβολικές και πρέπει να ομολογήσω ότι όλα αυτά είναι δυσχερέστατα να υλοποιηθούν. Μετά από πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου συστάθηκε μια άλλη ομάδα εκτός της Κομισιόν κάτω από την ηγεσία του κυρίου Στόιμπαρ. Και η Κομισιόν τώρα πρέπει να είναι σε θέση να μας πει ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση τέλος πάντων. Δηλαδή, ε, καλύτερη προσέγγιση της ομάδας της Κομισιό ή της εξωτερικής ομάδας που ε, ηγείται ο κύριος Στόιβερ. Ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση τέλος πάντων. Καμιά φορά υπάρχουν διάφορα επίπεδα ελέγχου στα κράτη-μέλη. Αναρωτιέμαι αν δεν θα μπορούσαμε να προσφύγουμε στην ιδιωτική βιομηχανία που έχει μεγάλες απαιτήσεις και θα μπορούσε να καταστήσει τους δημόσιους ελέγχους πλεονασματικούς. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τσινιάφσκι. Συμφωνώ με το ψήφισμα για την απλούστευση της ΚΑΦ. Της ΚΑΠ, με συγχωρείτε. Μπορείτε η Κομισιό να μας εξηγήσει τι ενέργειες έχουν αναλυφθεί ώστε να μειωθεί το διοικητικό βάρος για τους αγρότες μπορεί η Κομισιόν να μας ενημερώσει πώς σκοπεύει να δώσει συνέχεια στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωκοινοβουλίου για την απλούστευση. Πριν από τη μεταρρύθμιση, οι αγρότες ζητούν απλή πολιτική. Γιατί και στην Πολωνία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ευρύτερα υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις. Το έχουμε συζητήσει πολύ συχνά στο Ευρωκοινοβούλιο. Το συζητήσαμε και με την κυρία Άσουμποντ. Δεν μπορεί να μας καταστρέψει η γραφειοκρατία. η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αναπτυχθεί δεν μπορεί να δημιουργεί νέα εμπόδια ε, γραφειοκρατικά. Η κυρία Κίκαο τώρα. κάω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Η ΦΑΟ δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα ένα μνημόνιο στο οποίο λέει ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται εν ώψη νέων λίμων και ζητά να αυξηθεί η καλλιέργεια καλαμποκιού και σιταριού και ζητά να αυξηθούν τα αποθέματα ούτως ώστε να υπάρχει αυτάρκεια για περισσότερους μήνες. Πρέπει λοιπόν να ικανοποιήσουμε την παγκόσμια ζήτηση σε τρόφιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει όχι μόνο να διατηρήσει την παραγωγική της ικανότητα αλλά και να τη βελτιώσει. Θα πρέπει να ενισχύσει τις μικρομεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις όχι μόνο για τις άμεσες πληρωμές αλλά και για τις επιδοτήσεις. Εμείς θα πρέπει να τραβήξουμε στην αγορά τα προϊόντα από αυτές τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Οι γεωργοί χρειάζονται απόλυτη απλούστευση της γραφειοκρατίας. Θα πρέπει οι γεωργοί να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε χαμηλότοκα δάνεια. Σας παρακαλώ κύριε Επίτροπε για να μπορέσουμε να έχουμε επίσης και μειωμένο ΦΠΑ για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye και έχω να σας πω το εξής. Έχω εννέα αιτήσει, θα μπορούσα να δεχθώ πέντε. Θα καλέσω και τους εννέα, αλλά παρακαλώ να μην ξεπεράσετε ένα λεπτό για να μπορέσουμε κάποια ώρα να πάμε σπίτια μας απόψε. Ο κύριος Καλανόφσκι πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Κύριε Επίτροπε, στην ανακοίνωση της Επιτροπής η απλούστευση της ΚΑΠΑ επικεντρώνεται κυρίως στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Αυτή η πρόταση ουσιαστικά ακολουθεί τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχονται στο ψήφισμα του προηγούμενου Μαΐου. Η μείωση της γραφειοκρατίας θα επιτρέψει στους ε, γιοργούς να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πιο άνετη πληροφόρηση και θα υπάρχει και καλύτερος έλεγχος. Θα έχουμε λοιπόν ε, πιο ασφαλή προϊόντα και θα έχουμε και ασφάλεια στην αγορά. Πρέπει όμως η απλούστευση να είναι πραγματική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να εγγυθούμε ότι αυτές οι νέες προτάσεις δεν θα αποτελούν μία εξειδανικοποίηση ε, της πραγματικότητας. Πρέπει να μειώσουμε πραγματικά τη γραφειοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να μιλάμε για την γραφειοκρατία, γιατί ελπίζω ότι δεν θα είναι ε, εις βάρος μας. Χαίρομαι ε, κύριε Επίτροπε που πρεσβεύεται μία ε, απλοποίηση της γραφειοκρατίας για τις μικρές επιχειρήσεις και αυτό πρέπει να το επενέσουμε Καλό θα ήταν βέβαια να μην χρειάζεται κάθε ε, χρόνο οι γεωργοί να χρειάζουν ε, άδειε για τις ίδιες ε, εκτάσεις αλλά εάν δεν απλοποιήσουμε την γραφειοκρατία δεν θα επιτύχουμε τον τελικό μας στόχο και γι' αυτό αυτό το οποίο επιζητούμε ουσιαστικά θα είναι μια κοινή γεωργική πολιτική με λουλούδια στα χωράφια και όχι με χαρτιά στα γραφεία. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ανακοίνωση των γενικών αρχών σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να απλουστεύσουμε την ΚΑΠ δημιούργησε νέες ελπίδες στους Ευρωπαίους γεωργούς. Πρόκειται λοιπόν για τη διασφάλιση του ιδίου το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Χρειάζεται ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας. Οι γεωργοί δεν έχουν το χρόνο να αφιερώνονται σε διοικητικά ζητήματα χρειάζεται λιγότερος χρόνος και λιγότερο κόστος για τη γραφειοκρατία. Αν καταφέρουμε κάτι τέτοιο, θα έχουμε ένα σύστημα που θα μας οδηγήσει σε οικονομίες. Αξίζει τον κόπο κύριε Επίτροπε να το προσπαθήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση. Κυρία Μακίνε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για μια αυθεντική έκφραση της επιθυμίας του να προχωρήσει στην απλούστευση. Βεβαίως κανένας αγρότης δεν μου ζήτησε απλούστευση της ΚΑΠ. Ζήτησε λιγότερους ελέγχους και ευκολότερους τρόπους επιχειρησιακούς. Αλλά αν ακολουθήσουμε το δρόμο της ε, πρασίνησης του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ θα ενισχύσουμε την πολλαπλή συμμόρφωση, θα οδηγήσουμε περισσότερους στα, σε εκμεταλλεύσεις και δεν θα μπορέσουμε να πλουστεύσουμε, θα περάσουμε σε πράσινη γραφειοκρατία αντί σε κόκκινη γραφειοκρατία. Λοιπόν, ας έχουμε συνείδηση αυτού του θέματος. Υπάρχει και θέμα αξιοπιστίας. Οι τραπεζίτες στην Ευρώπη τα γλιτώνουν όλα Εκείνοι οι αγρότες δηλαδή συλλαμβάνονται για 100 ευρώ. Λοιπόν, οι αρμόδιες αρχές έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα φόβου. Εσείς φοβόσαστε κύριε Επιτροπέ τον προϋπολογισμό και οι αγρότες φοβούνται και τον τελευταίο επιθεωρητή. Πρέπει να σπάσει ο πόλεμος του φόβου. Ο κύριος Κυρσκεύσκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η διαχείριση του συστήματος ελέγχου και η διοίκηση είναι ένα φορτίο για τους προϋπολογισμούς των, κρατών. Βάσει της εμπειρίας μας μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα περίπλοκα κριτήρια για πρόσβαση σε ενίσχυση και όλοι οι έλεγχοι τελικά οδηγούν σε προβλήματα για τους αγιοργούς, αλλά και για την εθνική διοίκηση. Η ΚΑΠ πρέπει να είναι κατανοητή στους γεωργούς και στους φορολογούμενους. Χωρίς απλούστευση αυτό είναι ανέφικτο πια. Κάθε φορά που προσπαθήσαμε να μεταρρυθμίσουμε την ΚΑΠ, προσθέτουμε ουσιαστικά κι άλλο ένα στρώμα γραφειοκρατίας. Κάνω έκκληση λοιπόν στα κράτη-μέλη να μην προσθέσουν κι άλλες απαιτήσει μελλοντικά. Προτείνω ουσιαστικά για το μέλλον η αίτηση να καλύπτει ολόκληρη την περίοδο ενισχύσεων ετή με δυνατότητα τροποποίηση σε περίπτωση αλλαγών. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, από την ε, κοινή γεωργική πολιτική καταλήξαμε σε ένα περίπλοκο μηχανισμό ελέγχων ε, και πέρασε η γεωργία από τους αγρούς στα γραφεία των ε, υπαλλήλων στις Βρυξέλλες. Όλο αυτό το σύστημα εξαρτάται από τις επιδοτήσεις, πράγμα όμως το οποίο εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και η αγορά των τροφίμων ε, παρουσιάζει δυσκολίες ιδίως για τα νέα κράτη-μέλη διότι έχουν περιορισμένες δυνατότητες και γι' αυτό θα πρέπει να προσαρμοστούν τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να υπάρχει μία δίκαιη ρύθμιση για όλους και είμαι βέβαιος κύριε Επίτροπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας βοηθήσει σε αυτό το έργο. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ. Συμφωνώ πλήρως με την πρόταση αυτή να απλοποιήσουμε την κοινή γεωργική πολιτική και συμφωνώ απολύτως και με τον Επίτροπο και όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα διότι θα πρέπει καλύτερα να βασιζόμαστε στην εμπιστοσύνη και όχι στις κυρώσεις διότι οι γεωργοί νοιάζονται περισσότερο για τα χωράφια τους από ότι αυτοί οι οποίοι τους επιτηρούν και ε, δεν ε, θέλουν ούτε να χρησιμοποιούν υπερβολικά λοιπάσματα ούτε να μην κάνουν κάτι προς είτε της γης τους είτε των ε, ζώων αυτό που δεν θέλουν είναι να χρησιμοποιούν ε, ε, έγγραφα και αν το επιτύχουμε θα είναι προς όφελος όλων. Ο κύριος Λαβία. Κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, κάθε χρόνο το ελεγκτικό συνέδριο καταδεικνύει ότι όχι πάντα τα κονδύλια της ε, ΚΑΠ ε, χρησιμοποιούνται σωστά και διαφανώς. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να συνδυάσουμε δύο διαφορετικές απαιτήσεις. Δηλαδή αφενός την ανάγκη ελέγχου για να εγγυθούμε ότι οι φόροι των Ευρωπαίων φορολογουμένων χρησιμοποιούνται σωστά και από την άλλη να απλουστεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη ζωή των αγροτών μας οι οποίοι θέλουν να αφιερωθούν και είτε στην κτηνοτροφία είτε στην καλλιέργεια των χωραφιών τους. Εγώ θα ήθελα να πω στον Επίτροπο το εξής. Ε, όλα τα μέτρα, ε, τα ευρωπαϊκά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται μετά είτε από τα εθνικά κράτη είτε από τις περιφέρειες δεν απλουστεύουν καθόλου τα πράγματα πολλές φορές προσθέτουν γραφειοκρατία. Οι best practice, οι καλύτερες πρακτικές των ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών θα πρέπει να εφαρμόζονται γενικά. Ο κύριος Στογιάνοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ό,τι και να κάνατε μέχρι τώρα δεν ήταν επαρκές διότι διαφορετικά θα συζητούσαμε άλλα θέματα απόψε πρέπει να συζητήσουμε την κοινωνική πτυχή γιατί όταν κάποιος ετοιμάζει ένα, ε, ε, ε, να πάρει ένα δάνειο ετοιμάζει το φάκελό του αλλά μετά τα άτομα αυτά έχουν χροκοπήσει διότι εδώ και έξι μήνες προσπαθώ να διαπραγματευθώ με το Γεωργικό Ταμείο της Βουλγαρίας που απέριψε μία ολόκληρη σειρά προ προγραμμάτων και όπως ξέρετε η Βουλγαρία είναι υπό επιτήρηση οπότε προτιμά να απορρίπτει τα προγράμματα παρά να ε, οδύρεται αργότερα. Χρειάζονται πολλοί έλεγχοι. Έλεγχοι όμως αυτοί δεν πρέπει να αφαιρέσουν το ψωμί από το στόμα αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ ο κύριος Επίτροπος. Χωρίς μικρόφωνο. Oui. Donc, d'un côté, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχή από τη μια να βλέπω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος στην αίθουσα για να συζητήσει την απλούστευση τέτοια προχωρημένη ώρα. Νομίζω ότι εμείς είμαστε σαφείς όταν κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε, δηλαδή Υπάρχουν κανονισμοί, διατάξει είναι προτάσεις που έρχονται από την Κομισιόν, που περνάνε από το Συμβούλιο και περνάνε και από το Κοινοβούλιο. Ευελπιστώ λοιπόν ότι όταν εμείς θα επεξεργαστούμε από κοινού το νομοθετικό πακέτο, θα ξέρουμε σαφώς το τι θέλουμε και θα αποφύγουμε να προχωρήσουμε με εξαιρέσεις ή προσθήκες που μετά ερμηνεύονται με επιπλέον αρμοδιότητες της Κομισιόν για ελεγκτικού χαρακτήρα διότι η Κομισιόν μετά είναι υπόλογη σε εσά στο Κοινοβούλιο για τη σωστή χρήση του δημοσίου χρήματος. Η ΚΑΠ δεν εμποδίζει τους αγρότες να εργαστούν. Σε πολλές χώρες η ΚΑΠ είναι αυτή που βοηθάει τους γεωργούς να εργαστούν. Απλώς όταν πρόκειται για δημόσιο χρήμα ο καθένας θα πρέπει να έχει τη συνέστηση για το πώς το χρησιμοποιεί. Στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχουμε διατάξεις ειδικέ για το γεωργικό τομέα. Και πρόκειται για ε, έναν από τους εξαιρετικούς τομείς για τον στον οποίο γίνονται έλεγχοι επιτόπου για τη χρήση των κονδυλίων. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι. Η, εθνική, η ευρωπαϊκή λοιπόν νομοθεσία απαιτεί επιτόπου έλεγχο. Αυτό το οποίο θεωρείται πολύπλοκο είναι όλη η νομοθεσία για το περιβάλλον, για την ευημερία των ζώων. Είναι διαδικασίες για ορισμένα ειδικά μέτρα όπως είναι τα μέτρα για την οικοσυμβατότητα όπως επίσης και τα μέτρα επένδυσης που τα έχουμε στα προγράμματα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Η νομοθεσία στην πράξη, έτσι όπως ερμηνεύεται στην πράξη, πρέπει να βελτιωθεί αλλά για τις διαδικασίες, για τα ειδικά μέτρα, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιομορφίες της κάθε περιφέρειας και χρειάζονται και αντίστοιχη έλεγχοι γιατί αλλιώς δεν είμαστε αξιόπιστοι. Σύμφωνο ότι πρέπει να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο με την απλούστευση. Αλλά δεν θέλω να προχωρήσουμε πια τόσο πολύ, ούτως ώστε να καταστούμε αναξιόπιστοι ως προς τη διαχείριση του χρήματος της ΚΑΠ. Θα ήθελα πάντα ο προϋπολογισμός για την ΚΑΠ να παραμείνει παχυλός στο μέλλον. Και για να παραμείνει εξίσου υψηλός αυτός ο προϋπολογισμός θα πρέπει να ξέρουμε πώς χρησιμοποιείται. Τώρα για τη διαφάνεια υπάρχει μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εγώ ε, λαμβάνω υπόψη μου την απόφαση του δικαστηρίου και τον σχετικό κανονισμό για την διαφάνεια. Θα τελειώσω εδώ. Ε, θα σταματήσω εδώ το λόγο μου, αλλά δεν θα σταματήσω όμως τη δράση μου για να προχωρήσω στην απλούστευση της ΚΑΠ. Επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά ότι θα πρέπει η δουλειά να είναι καρπός συνεργασίας μεταξύ ημών και των κρατών μελών. Γιατί εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε στη μείωση της γραφειοκρατίας ως προς αυτά τα οποία θα ζητάει η Κομισιόν στα κράτη-μέλη, αλλά την ευθύνη για τη διαχείριση της ΚΑΠΤΑ έχουν τα κράτη-μέλη. Οπότε το πρόβλημα της γραφειοκρατίας πολλές φορές έχει να κάνει με το πώς ερμηνεύονται οι κανονισμοί από τα κράτη-μέλη και από τις περιφέρειες. Σίγουρα θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτούς τους οδηγούς των καλύτερων πρακτικών, αλλά σήμερα με την συναπόφαση έχετε ε, τις ίδιες αρμοδιότητες με το Συμβούλιο και είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έληξε η συζήτηση και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα μας. Η προφορική ερώτηση που αφορά την κατάσταση στο μελισσοκομικό τομέα. Ο κύριος Δεκάστρο έχει πέντε λεπτά.